Θα ξεκινήσουμε αμέσως με το επόμενο σημείο της εμερήσιας διάταξης γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Στην ημερήσια διάταξη, I'm assuming that the Commission speaks Greek because you don't have your things on. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την κατάσταση στην Ουκρανία. Με δεδομένο ότι δεν μπορεί να είναι παρούσα, την Επιτροπή εκπροσωπεί ο κύριος Φούλε. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Thank you uh, Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής η κάθε άστον μου ζήτησε να προβώ στα κάτω τη σχόλια.